Ε, αποδέκτες. Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνει εδώ μια ε, μακρά χρονιά. Σας ε, ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Καλή επάνωδο στα σπίτια.